για άρνηση της, ε, του να δοθεί η συγκατάθεση και 174 υπέρ της. Η, η είναι η κυρία Βαλενσιανό. Θα γίνει συζήτηση για 25 τροπολογίες. Δίνω το λόγο στην συγγήτρια η οποία θα μας εκθέσει τις δικές απόψεις σχετικά με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Κυρία Βαλενσιάνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Λαμπρινή και τον κύριο Σέφερ, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την οριστική συζήτηση στην Επιτροπή για την Συμφωνία Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας με την Κούβα. Θα μιλήσουμε κυρίως για το ψήφισμα που συνοδεύει την συνένεση του Κοινοβουλίου και που δέχτηκε τις περισσότερες ε, ε, τροποποίησης. Δεν χρειαζόταν, δεν ήταν απολύτω απαραίτητο, αλλά αυτό που αποφάσισε η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών. Ως εισηγήτρια προετοίμασα ένα ψήφισμα το οποίο θεωρώ ισορροπημένο και που μιλά για την πολιτική συμφωνία και όχι για την πολιτική κατάσταση της Κούβας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ψήφισμα συνοδεύει την ε, ε σύμφωνη γνώμη μας για την πολιτική συμφωνία και δεν σχολιάζουμε την πολιτική κατάσταση στην Κούβα. Το επιμένω γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για την συνεισφορά τους. 274 τροπολογίες ε, κατέθηκαν, 66 από το ΕΛΚ, 42 από τους φιλελεύθερους κλπ. 81 συμπεριλήφθησαν στις 25 συμβαστικές προτάσεις που προετοίμασα. Άλλες 21 θα υποστηριχθούν από την συγκεκριμένη από την υποφαινόμενη, συνολικά 102, δηλαδή το 56% των κατατεθειμένων μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ε, συμπεριλήφθησαν ή θα υποστηριχθούν. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι το ποσοστό ή το απόλυτο νούμερο, αλλά το περιεχόμενό τους. Προσπάθησα να καθησυχάσω και να λάβω υπόψη μου τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα όλων σε ένα ζήτημα το οποίο είναι περίπλοκο με θέσεις ε, πολύ, που πολύ απέχουν μία από την άλλη συχνά. Προσπαθώ όμως παρόλα αυτά να εξασφαλίσω τη μέγιστη δυνατή συνένεση ώστε η έκθεση να είναι λογικά συνεπής και βέβαια γι' αυτό το λόγο όλοι χρειάζεται να κάνουμε και θυσίες και παραχωρήσεις. Στις 17 έλαβε χώρα η δεύτερη συνάντηση των σκιωτών εισηγητών και αφού ε, αναλύσαμε τις ε, συμβαστικές προτάσεις ε, που είχα καταθέσει, κάποιοι συναδελφοί από τους φιλελεύθερους και από το ΕΛΚ ζήτησαν να συμπεριφθούν καινούρια στοιχεία. Τους ζήτησα Ζήτησα από τους κοιόδης ηγητές να μου στείλουν τα σχόλιά τους. Η συνάδελφος των φιλελευθέρων μου τα έστειλε, την ευχαριστώ δημοσίως για την δουλειά της. Όμως θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που είπα και στην συνάντηση των σκιωδών ηγητών. Το έχω πει επανειλημμένος άλλωστε. Για να δεχτώ ή να απορρίψω τις τροπολογίες χρησιμοποίησα συγκεκριμένα κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι αυτό που είπα στην εισαγωγή. Μιλάμε για ένα ψήφισμα που συνοδεύει μια σύμφωνη γνώμη για την Συμφωνία Πολιτικού Διαλόγου και Συνασίας με την Κούβα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία λοιπόν αποκλείονται από την, ε, το ψήφισμα. Δεύτερον, ε, πέριψα λεπτομερείς περιγραφές της κατάστασης στην Κούβα. Γιατί και πάλι αυτό διαφεύγει του ψηφίσματος. Επίσης αρνήθηκα να αναφερθώ σε συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει και το κάναμε να συζητήσουμε με τον κύριο Λαμπρινίδη. Με τον κύριο Λαμπρινίδη θα πρέπει να εμπεδώσουμε ένα σύστημα παρακολούθηση του διαλόγου σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα με την κουβανέζικη κυβέρνηση. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να παρακολουθούμε την πρόοδο που θα λαμβάνει η ενδεχομένω χώρα, αλλά δεν νομίζω ότι το ψήφισμα θα πρέπει να αναφέρεται σε μεμονωμένε περιπτώσει, χωρί αυτό να σημαίνει ότι οι μεμονωμένε περιπτώσει δεν είναι σημαντικέ και δεν μα απασχολούν. Απλά δεν είναι, δεν εμπίπτουν οι μεμονωμένε περιπτώσει στο πεδίο του ψηφίσματος. Από την οπτική γωνία της δικής μου πολιτικής ομάδας, οι, οι δεσμεύσεις οι οποίες αναλαμβάνουμε είναι σαφείς. Αλλά η δική μου, ο δικός μου στόχος δεν ήταν να ε, προωθήσω την άποψη της δικής μου πολιτικής ομάδας. Προσπαθώ να βρω ένα κοινό παρανομαστή για όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι προφανές ότι η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων της Ευρωβουλής θέλουν να δουν αλλαγές στην Κούβα. Θέλουν μεταρρύθμιση του πολιτικού συστήματος στην Κούβα και θέλουν κυρίως μια βελτίωση της καθημερινής ζωής των Κουβάνων. Των Κουβανών. Αυτό είναι κοινό παρονομαστή σε όλες τις πολιτικέ ομάδε. Όχι. Ε, δεν, θέλουν όμως όλοι να επιλέξουν τον ίδιο δρόμο, το ίδιο μονοπάτι. Γι' αυτό το λόγο και εγώ πρέπει να κάνω κάποιε επιλογέ έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια πλειοψηφία. Επειδή όλοι θέλουμε να βελτιωθεί η κατάσταση στην Κούβα, όλοι θέλουν αυτό που ονομάζουν ε, μεταπολίτευση, εκδημοκρατισμό κλπ. Αλλά πιστεύω ότι το καλύτερο εργαλείο είναι ο πολιτικός διάλογος. Δεν βλέπω τι θα κερδίζαμε αν παρεμποδίζαμε αυτό τον διάλογο. Και με τη συμφωνία σίγουρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα για να γίνει ο πολιτικός διάλογος. Για να επικυρωθεί όμως μια συμφωνία χρειάζονται, χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών. Και από αυτή και από την άλλη μεριά του Ατλαντικού ωκεανού. Χωρί λοιπόν συμφωνία πολιτικού διαλόγου θα ήταν πολύ δύσκολο η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ τι αλλαγέ. Σίγουρα χωρίς αυτή τη συμφωνία η ισχύ μας θα είναι πολύ μικρότερη να επηρεάσουμε υπέρ των αλλαγών. Να σας πω ποιες είναι αυτές οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε. Από τις 25, 25 ε, συγγνώμη, συμβαστικές προτάσεις από τις 25 οι 8 αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από τις 25 συμβαστικές προτάσεις οι 8 αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα δείχνουμε στην Κούβα ποια είναι τα πρότυπα προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία θέλουμε να ε, δεχτεί, συμβαστική πρόταση 4 και 5, καθορίζουμε τις πολιτικές μας προτεραιότητες ό,τι αφορά τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τον, τον οικονομικό εξυγχρονισμό για τη βελτίωση της καθημερινότητας, αυτή είναι η συμβαστική πρόταση 8 και 24, στην 11 Μιλάμε ξανά για τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ελευθερία έκφρασης, ε, συνεταιρισμού και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και για την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και άλλων πολιτικών φορέων χωρίς περιορισμούς. Ζητούμε επίσης εγγύησεις για το, την, ε, την εργασία των ε, υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην συμβαστική πρόταση 13 πάλι μιλάμε για τις ελευθερίες και, τις και για τα πολιτικά δικαιώματα. Στις 15, στις 15 και την 20 μιλούμε πάλι για τη συμμετοχή τη κοινωνίας των πολιτών και της ελευθερίας. Στην 22 δε μιλούμε για, πάλι για την ανησυχία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, βλέπετε ότι ε, δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην, στις που υπάρχουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και συγκεκριμένους στόχους. Στην συμβαστική πρόταση 9 μιλάμε για πολιτική μεταρρύθμιση, πολιτική και οικονομική μετάβαση, χρήση των εργαλείων της εξωτερικής πολιτικής για να ενισχυθεί ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών που στηρίζει μια ειρηνική μετάβαση και θα ήθελα οι συνάδελφοι να ε, αξιολογήσουν σωστά το κείμενο αυτό. Μιλάμε για μετάβαση δημοκρατική, μετάβαση εκδημοκρατισμό δηλαδή. Δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να πάμε πιο μακριά από αυτό. Στην συμβαστική πρόταση 10 λέμε ότι οι δεσμεύσεις ε, οι υποχρεώσεις είναι δεσμευτικές και για τις δύο πλευρές. Ε, καταγγέλουμε το εμπάργκο και την εφαρμογή της εξοδικαστικής νομοθεσίας ε, στη 17 και την 20. Στη 14 και την 23 μιλούμε για την, οικονομική, το οικονομικό άνοιγμα και τις εγγύησεις στη 16. Μιλάμε για την αντιπροσωπεία που έχουμε αποφασίσει να στείλει το κοινοβούλιο. Ε, έχει γίνει δεκτή, δεκτό το ταξίδι, αλλά όχι η ημερομηνία ακόμα. Στο συμβαστική πρόταση 12, παρακαλώ πολύ προσοχή εδώ, γιατί πιστεύω ότι δεν θα αρέσει καθόλου στις κουβανίζικες αρχές, μιλούμε για ειδική λογοδοσία από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων προς το Κοινοβούλιο προκειμένου να παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί, γιατί είναι μια συμφωνία ιδιαίτερης πολιτικής ευαισθησίας. Νομίζω ότι υπάρχει μια ευρεία συνένεση υπέρ αυτής της συμφωνίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Η ίδια συνένεση υφίσταται και μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό συνέβαινε και πριν από 20 χρόνια Ενώ η κοινή θέση λειτουργούσε και είχαμε και 22 κράτη-μέλη είχαν υπογράψει πάνω από 90 διμερείς συμφωνίες με την Κούβα. Και λέω αυτό κατά τη διάρκεια της περίοδου που υφίστατο η κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ζητώ, το λέω για να ζητήσω από τους να στηρίξουν τις συμβαστικές προτάσεις. Νομίζω ότι είναι η βάση, η μέγιστη βάση, ο μέγιστος κοινό πανομαστής τον οποίο μπορούμε να βρούμε. Είναι σημαντικό το ψήφισμα να διατηρήσει την λογική του συνοχή. Δεν είναι δυνατό με το ένα χέρι να ανοίγουμε την πόρτα και με το άλλο να την κλείνουμε. Θέλουμε ένα διάλογο με την Κούβα που θα βασίζεται σε ισχυρέ απαιτήσει σε ό,τι αφορά τις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα διάλογος ο οποίος να έχει αυτά αποτελέσματα που να μπορεί να τα αξιολογήσει και να τα μετρήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά και περιμένω να ακούσω και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αβάνα ε, περιμένει την απόφαση αυτή και του έχω υποσχεθεί ότι θα βρούμε τον καλύτερο δυνατό δρόμο που είναι πράγματι η οδός που θα οδηγήσουν τους κουβανούς και τους κουβανές σε ένα, ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στους ε, σκιώδεις εκ μέρους του ΕΛΚ, ο πρώτος ε, σκιώδης ομιλητής. Ζητώ συγγνώμη γιατί τα, το αεροπλάνο μου καθυστέρησε και δεν κατάφερα να παραστώ στην ε, παρουσίαση του κυρίου Λαμπρινίδη. Ζητώ συγγνώμη. Φαντάζομαι ότι δεν θα αμέλησε να παρουσιάσει κάποιες πτυχές της κατάστασης στην Κούβα. Ε, ζητώ συγγνώμη λοιπόν που δεν ήμουν παρόν. Θα μιλήσω εκ μέρους του ΕΛΚ, Γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα και ο εξή περιπλοκο ήταν και ο ρόλος της ηγητρίας. Είναι άνθρωπος μετρημένος, ε, είναι άνθρωπος ισορροπημένος, προσπαθεί να βρει ισορροπίες ε, όλοι θέλουμε να είναι ισορροπημένοι η, η νομοδότηση. Βέβαια, ε, οι, οι τεχνικοί κανόνες επιτρέπουν να συνοδεύεται κάπου ένα ψήφισμα και εκεί περιπλέκονται τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι θα στηρίξουμε τη σύμφωνη γνώμη. Ε, όχι για να επενέσουμε την κουβανέζικη πλευρά που δεν έχει κάνει πολλά πράγματα, αλλά για λόγους ιστορικής συγκυρίας και ιστορικών απαιτήσεων. Όπως λέει και η συγκυτρία θα πρέπει να προσπαθήσουμε δεχομένω να σιωπήσουμε κάποια λόγια τα οποία θα θέλαμε να προφέρουμε, ε, αλλά που θα ήταν ε, άκερο να εκφραστούν αυτή τη στιγμή. Θα κάνω λοιπόν μια προσπάθεια και εγώ ίδιος και θα προσπαθήσω η ομάδα μου να ε, συμμορφωθεί με την βασική συμφωνία την οποία προτείνεται μέσω των συμβαστικών προτάσεών σας. Ευχαριστούμε πολύ που υποβάλλατε αυτές τις συμβαστικές προτάσεις. Ε, προσπαθείτε να ικανοποιήσετε πολλές από τις ανησυχίες που εξέφρασαν και άλλες πολιτικές ομάδες, όχι μόνο η δική μας. θα πρέπει ε, να κάνουμε προσπάθεια να υποχωρήσουμε, παρόλο που δεν ικανοποιούμαστε πλήρως, ακριβώς εξαιτία της ιστορικής σημασίας της στιγμής. Ε, η... Πρέπει να αν αντιληφθούμε ότι η Κούβα έχει κάνει ε, δρόμο, πολύ ανεπαρκή βέβαια, αλλά θα πρέπει να το ε, αναγνωρίσουμε. Θα ε, μελετήσουμε τις σημαντικές προτάσεις. Αν έχουμε να κάνουμε κάποια, αν έχουν κάποιο αίτημα βελτίωσης, θα το επιβάλλουμε γραπτός θέλουμε ε, να πούμε ότι πολλά μέλη της ομάδας μας έχουν θεμητές αντιρρήσεις, θεμητές επιφυλάξεις και θα ήθελα να επιφυλαχθώ και εγώ να μελετήσω καλύτερα τις συμβαστικές προτάσεις. Κάποιοι από τους συναδέλφους της ομάδας μου είναι πιο απαιτητικοί από μένα και ενδεχομένως θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε προς αυτήν την κατεύθυνση, κυρία Συγκήτρια, κάποια πρόσθετη συμβαστική πρόταση για να καλυφθούν και αυτοί. Ξέρω ότι κάποια πράγματα είναι δύσκολο να ληφθούν, αλλά είναι αδύνατο να μιλήσουμε για την Κούβα και να μιλάμε για, τα, για τους πολιτικούς κρατουμένους. Είναι αδύνατον να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά όταν ε, ε, άτομα τα οποία έχουν λάβει το βραβείο Ζαχάροφ ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μα ζητούν να μην υπογράψουμε συμφωνία και εμεί θα την υπογράψουμε παρόλα αυτά. Ε, και ζητώντα του συγγνώμη γιατί έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο που μα ζητούν να μην προβούμε σε τέτοια συμφωνία, αλλά πολλέ φορέ η πολιτική είναι η τέχνη του δυνατού. Οπότε θα σας ζητήσουμε κάποιες ακόμα συμβαστικές προτάσεις. Πιστεύω ότι θα βρούμε μια ένα κοινό πεδίο. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε για δύο-τρία πράγματα ακόμα. Ε, από το ψήφισμα όλοι περιμένουν να ζητήσουν από την Κομισιόν ένα ε, οδικό χάρτη διαφανή και απτό αυτό όμως που δεν ζητούμε καθόλου στις προτάσεις είναι η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Τελειώνω, Πρόεδρε. Ο Ραούλ Κάστρο ε, ρώτησε, ε, μάλλον ένας δημοσιογράφος ε, ρω, ε, ρώτησε τον ε, Ραούλ Κάστρο για τους πολιτικούς κρατούμενους και είπε ο Ραούλ Κάστρο πέστε μου ποιοι είναι να τους απελευθερώσω αύριο. λες και δεν τους ξέρει το σύστημα, το καθεστώς. ...432 αυθαίρετες συλλήψεις ε, έχουν επιβεβαιωθεί από, τον, από την ε, Κουβανέζικη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν θα επιμείνω σε αυτό το θέμα. Ε, κάποιοι συνάδελφοι στην ομάδα μου έχουν διαφορετική άποψη από μένα, είναι πιο απαιτητικοί, ε, ζητούν στο ψήφισμα να αναφερθούν όλες οι ανησυχίες τους και πιστεύω ότι θα πρέπει να υποφεληθούμε τις ευκαιρίες του ψηφίσματος και να τα αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι εγώ, είμαι ο επόμενο ομιλητή, ο υποφαινόμενο, γιατί εκπροσωπώ το κόμμα ΙΣΙΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά σα, για τη συνεργασία. Όπω έχω πει επανειλημμένα, είμαστε ανοιχτοί, αλλά παράλληλα θεωρούμε ότι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι το πιο σημαντικό σε αυτό το διάλογο, γιατί δεν βλέπουμε να υπάρχουν οικονομικοί, πολιτιστικοί και άλλοι παράγοντε που να είναι πιο σημαντικοί στη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση-Κούβα. Και γι' αυτό εμεί κόμμα, πολιτική ομάδα έχουμε καταθέσει τροπολογίες και εγώ και κάποια άλλη από την ομάδα μου θα χαιρόμασταν πάρα πολύ αν ε, τις δεχτείτε Τις δεχτήκατε κάποιες στους συμβασμούς, άλλες πάλι όχι. Εμείς θα ασκήσουμε ακόμα μεγαλύτερη πίεση για να υπάρχει ισορροπία στις δύο εκθέσεις. Στη τελική ανάλυση αυτό είναι ο στόχος ε, της πολιτικής μας ομάδας. Και προσβλέπουμε στη συνεργασία και ελπίζουμε τελικά να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ε, συμβαστική πρόταση όπου θα μπορέσουμε και να ε, στηρίξουμε το τελικό αποτέλεσμα της έκθεσης. Αυτά εκ μέρους της ε, πολιτικής μας ε, ομάδας. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στην σφιλέτερη, στην κυρία Μίκινες. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια κύριε Βαλενθιάνο. Είμαι σίγουρη ότι κάνετε ό,τι μπορείτε. Προσπαθείτε να δείξετε όσο μεγαλύτερη ευελιξία γίνεται για να μας ικανοποιήσετε όλους. Νομίζω ότι σίγουρα βαίνουμε προς μια συμφωνία. Θα δουλέψουμε τις συμβαστικές προτάσεις. Ε, το σημαντικό είναι όμως να μην μείνουν εκτός σημαντικά θέματα τα οποία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Θέλουμε να είμαστε όσο πιο αυστηροί γίνεται, μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο βέβαια. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα προδώσουμε τους κουβανέζους φίλους μας που μας παρακολουθούν από πολύ κοντά. Για παράδειγμα, ε, τους ανθρώπους στους οποίους απονεμήθηκε το βραβείο Ζαχάροφ. Εφόσον αποφασίσαμε να επεξεργαστούμε ένα ψήφισμα, είναι ευκαιρία να συμπεριλάβουμε ένα, μια σειρά ζητημάτων. Θέλουμε αυτό το ψήφισμα να αποτελέσει, να βρίσκεται στη μεριά των κουβανίζων πολιτών και όχι στη μεριά της δικτατορίας. Πιστεύω ότι τελικά θα συμφωνήσουμε. Θα διαπραγματευτούμε όπως κάναμε πάντοτε και με σίγουρο θα βρούμε ένα σημείο σύγκλησης. Ευχαριστώ. Thank you, Όπως είπε και ο κύριος Δεγκράντες και εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη ε, που έφτασα καθυστερημένος και να επωφεληθώ για να επενέσω τον κύριο Λαμπρινίδη για την εξαίρετη δουλειά που κάνει στην Κούβα. Έχω μιλήσει και διμερός από κοντά μαζί του. Θέλω να το κάνω και δημοσίως ε, ο διαρθρωμένος διάλογος αυτή τη στιγμή γίνεται σε συνθήκες που δεν είχε γίνει ποτέ στα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό να τον ακούσουμε λοιπόν και να τον ευχαριστήσουμε. Την άλλη μεριά δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που έχουμε πει σε παλαιότερες συζητήσεις. Εκ μέρους της ομάδας μας θέλω να πω ότι οι συμβαστικές προτάσεις της ηγήτριας είναι σημαντικές αξιόλογες ε, τις ε, αξιολογούμε αυτή τη στιγμή. Επιμένουμε ότι μια καινούργια σχέση με το νησί θα πρέπει να συνοδεύεται προφανώς από μια πολύ πλειοψηφική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, η ομάδα μου θέλει η, συνένεση αυτή να εξασφαλίσει, η συμφωνία αυτή να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη τη συνένεση. Θα ήταν όμως πολύ κακό να να δώσουμε μια σύμφωνη γνώμη στην ε, συμφωνία. Και κατόπιν το ψήφισμα το οποίο την ακολουθεί να αντιτίθεται κάθετα στην δεκτικότητα της ε, κουβανέτικης πλευράς. Προφανώς μας ανησυχεί το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, αλλά 8 από τις 25 συμβαστικές προτάσεις αναφέρονται σε αυτό το ζήτημα. Ποιο άλλο, ποια άλλη έκθεση για χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση συνάπτει κάποια συμφωνία, έχει συνάψει κάποια συμφωνία, κάνει τόσες πολλές αναφορές όσο αυτή στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ δε περισσότερο θα είχα ανησυχίες αν γινόταν προσπάθεια να γίνει ακόμα πιο αυστηρό το κείμενο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υποσκάπταμε την συνένεση για τη συμφωνία. Μην ξεχνάμε ότι και η Κομισιόν και πολλά κράτη-μέλη ήδη εργάζονται ε, στη σύσφυξη των σχέσεων με την Κούβα. Πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, έχουν ήδη προγραμματίσει επισκέψεις στο νησί και δεν πιστεύω ότι θα ήταν σωστό να παρεμποδίσουμε με κάποιο τρόπο αυτές τις επισκέψεις, αυτή τη σύσφυξη των σχέσεων ε, από πλευρά διαφόρων κρατών μελών με την ΚΟΠΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ούτεσουν. Ο κύριος Αλαφράγκα. Ο κύριος Τεγράντες εξήγησε πολύ καλά την θέση της πολιτικής ομάδας. 27 κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο οι υπηρεσίες εξωτερικής δράσης και η Κομισιόν ζήτησαν από το Κοινοβούλιο να δώσει την σύμφωνη γνώμη του. Σε ό,τι αφορά τη δική μας πολιτική ομάδα, δεν θεωρώ ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα στην έγκριση, στην έγκριση της συμφωνίας. Τώρα που και πέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του, μια γνώμη που δεν απαραίτητο θα πρέπει να έχει ως στόχο να ικανοποιήσει, να χαροποιήσει την, την κουβανέζικη κυβέρνηση. Όπως μας εξήγησε ο ειδικό εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, η Κούβα δεν είναι η αρχαία Αρκαδία, ε, ο παράδεισος επί της γης. Ε, εγώ δεν θα ζητούσα από την Κούβα κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουμε ζητήσει σε, από άλλες χώρες, όπως η Κολομβία για παράδειγμα στη Λατινική Αμερική. Θα ζητούσα λοιπόν από την εισηγήτρια, δεδομένου ότι έχω υπογράψει κάποιες τροπολογίες, να κινητοποιήσει ακόμα περισσότερο την καλή της θέληση, προκειμένου να μας ικανοποιήσει λίγο περισσότερο έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να πάρει μια σαφή στάση. Κανείς, όπως είπε ο κ. Τεγκράντες, δεν θέλει να εμποδίσει την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας, αλλά σε κάθε περίπτωση η Κούβα είναι μια ανομαλία η οποία δεν είναι δική μας ευθύνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω. Κυρία Βαλεντιάνο, για τις καταληκτικές παρατηρήσεις σας παρακαλώ. Bueno, Προφανώς είμαι ανοιχτή να εξετάσω καινούριε προτάσεις. Έχω την εντύπωση όμως ότι έχω φτάσει στα όρια μου, στα όρια του της λογικής συνέπειας. Έτσι πρέπει να είμαστε λογικός συνεπείς. Κάποιοι λένε η συμφωνία δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά θα βάλουμε τόσες πολλές καταγγελίες ή προβλήματα στο κείμενο το οποίο τη συνοδεύει, που μου φαίνεται σαν να μην είναι να μην συμβαδίζουν αυτά τα δύο. Η συμφωνία είναι συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασία Δεν είναι εμπορική ε, συμφωνία κύριε Σαλαφράγκα, δεν μπορούμε να τα αναμίξουμε, το ξέρετε πολύ καλά. Είναι μια συμφωνία για να ξεκινήσουν αυτά τα οποία θέλουμε να ξεκινήσουμε με την Κούβα. Δεν είναι μια εμπορική συμφωνία η οποία πρέπει να απαιτεί συγκεκριμένους κανόνες, στάνταρ πρότυπα κλπ. Είναι μέσω του διαλόγου που θα γίνουν αυτές οι, θα γίνει αυτή η πρόοδος. Οπότε δεν έχει σχέση αυτή η συμφωνία με τις άλλες οποίες αναφέρατε. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι την τελευταία στιγμή θα διαπραγματευτούμε υπό την προπόθεση ότι θα εξακολουθούμε να είμαστε λογικά συνεπεί. Δηλαδή, αν συμφωνούμε να ανοίξουμε ένα, μια καινούργια σελίδα με την Κούβα, το κάνουμε. Και στο πλαίσιο αυτή τη καινούργια σελίδα, α εμπεδώσουμε αυτή την σχέση, α προσπαθήσουμε να ε, επηρεάσουμε, α υπερασπιστούμε τι αξίε μα κλπ. κλπ. Έτσι κι αλλιώ, όπω είπε και κάποιο συνάδελφο, Ήδη τα κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει σε αυτό τον πολύ πιο προχωρημένο διάλογο με την Κούβα. Και εμείς θα πρέπει να βασιζόμαστε και να λαμβάνουμε υπόψη την πραγματικότητα όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην Κούβα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Okay, gracias. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βαλεντιάνο. Στο τέλος της συζήτησης θέλω να πω ότι η ψηφοφορία θα γίνει στις 20 Ιουνίου στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και η τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει μάλλον τον Ιούλιο. Λοιπόν, μπορούμε τώρα να περάσουμε στα σημεία 8 και 9, συμφωνία με τη Νέα Ζηλανδία, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε, θα σταματήσουμε τώρα, θα διακόψουμε τη συνεδρίασή μα και θα επανέλθουμε εδώ στι 5, γιατί ο συγγητή μα, ο κύριο Τάνικ δεν είναι εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν στι 5 και ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον κύριο Σέφερ για την παρουσία του εδώ στην Επιτροπή μας. Υπότιτλοι στον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 We will resume the meeting with, um, Συνάδελφοι, συνεχίζουμε και θα δούμε τώρα τα σημεία. Το σημείο 7. Όχι, λάθος. Τα σημεία 8 και 9. Τα αλλάξαμε είπαμε. Συμφωνία εταιρική σχέση για τη σχέση και τη συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών τη αφενό και τη Νέα Ζηλανδία αφετέρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νέα Ζηλανδία δεσμεύονται να συνεχίσουν τις μακροχρόνιες σχέσεις τους και η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για τη Σχέση και τη Συνεργασία υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2016 που αποτελεί ένα μελλοντοστραφές πολιτικό πλαίσιο για τη σχέση μεταξύ των δύο μερών. Αφορά μια σειρά αποζητήματα, ανθρώπινα δικαιώματα, καταπολέμηση της δημοκρατίας, οικονομική συνεργασία, ε, κλιματική αλλαγή, συνεργασία σε ζητήματα επιστήμης και τεχνολογίας. Οι διαπραγματεύσεις ε, θα ξεκινήσουν ε, σύντομα. Ο Πρωθυπουργό Νέα Ζηλανδία επισκέφθηκε τι ε, Βρυξέλλε τον Ιανουάριο. Ε, Εντό του πρώτου μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων του, κάτι που αποτέλεσε και ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία που αποδίδει στη σχέση με, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Τάνοκ, τον συγητή μα, για την ε, σύσταση και την ε, έκθεση για την ε, συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Η Συμφωνία Εταιρική Σχέση για τη Σχέση και τη Συνεργασία που είναι γνωστή και ως ΠΑΡΚ μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νέας Ζηλανδίας είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη. Η Νέα Ζηλανδία είναι μια, είναι μια χώρα με την οποία μας συνδέουν κοινέ αξίες και αρχές. Και η ΠΑΡΚ ε, βασίζεται σε μια ε, συμφωνία που είχε συνεχθεί το 2007 πλέον και προέβλεπε στενή συνεργασία και διάλογο σε επίπεδο υπουργών. Τώρα πια λοιπόν έχουμε ένα σχέδιο ψηφίσματος με το οποίο επανεπιβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας στη συμφωνία και με το οποίο εκφράζουμε την βαθιά μας αλληλεγγύη με την Νέα Ζηλανδία. Η ΠΑΡΚ καλύπτει πολλούς τομείς και ε, είναι παρόμοια με την συμφωνία που υπεγράφει πρόσφατα με τον Καναδά, για την οποία ήμουν επίσης ηγητής. Μιλούμε για την καταπλήρωση της τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος, ε, παγκόσμια ανθρωπιστική βοήθεια, συνεργασία σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, αντιπετώπιση κλιματικής αλλαγής και υποστήριξη βιώσιμης ανάπτυξης. Η Νέα Ζηλανδία είναι ηγέτης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έχει θέσει φιλόδοξους στόχους ε, που είναι παρόμοιοι με εκείνους που έχουν θέσει πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης. Αυτό αφορά την καταπολέμηση της ε, κλιματικής αλλαγής, την υποστήριξη βιοποικιλότητας και αυτές οι αρχές ε, διαπνέουν ολόκληρη την ΠΑΡΚ, κάτι που υποστηρίζω. Το άρθρο 15 που αφορά την, συνεργασία για την εφαρμογή της συμφωνίας του ΠΟΕ για υγειονομικά και φυτο-υγειονομικά ζητήματα επίσης δίνει ε, μια αίσθηση για τη δέσμευση που, για τις δεσμεύσεις που έχουν λάβει και τα δύο μέλη. Επίσης η ΠΑΡΚ επιβεβαιώνει την ε, συμφωνία που είχε υπογραφεί το 2012 που επιτρέπει την Ζηλανδία να συνδράμει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αποστολές της ε, κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ε, αυτό δίνει τη δυνατότητα και στη Νέα Ζηλανδία να διαδραματίσει έναν παγκόσμιο ρόλο που είναι και ιδιαίτερος αν λάβει κανείς υπόψη του το, το μικρό μέγεθος και τον μικρό πληθυσμό αυτής της χώρας. Ε, αυτό ε, έγινε ιδιαίτερα εμφανές και στην συμβουλή που είχε η Νέα Ζηλανδία στην, στις αποστολές Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της πειρα, Επίσης, στο ψήφισμα αναδεικνύεται ο ρόλος που έχει ε, διαδραματίσει η Νέα στις ε, αποστολές αστυνόμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Μάλιστα, ε, κατά την σύνοδο με το Αφγανιστάν ήταν σημαντικό το στοιχείο το ότι είχε υπογραφεί η ΠΑΡΚ τον Οκτώβριο και νομίζω λέγον, ε, ότι μιλώ ε, εκ μέρους της πλειοψηφίας ότι είναι θετικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τηρήσει μια θετική στάση απέναντι στη Νέα Ζηλανδία γιατί η Νέα Ζηλανδία είναι μια δύναμη του καλού στον κόσμο. Ε, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες οι οποίες βελτιώνουν το κείμενο, ιδίως όσον αφορά την, την περιφερειακή συνεργασία. Ελπίζω οι περισσότερες τροπολογίες ε, να είναι ε, με παρόμοιο τρόπο επικοδομητικές. Συμπερασματικά νομίζω ότι η υπογραφή της ΠΑΡΚ δεν είναι απλώς μια θετική εξέλιξη σχέση Ένωσης και Νέας Ζηλανδίας, αλλά αποτελεί ένα τμήμα μιας ευρύτερης ε, διαδικασίας επιτυχιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις συμφωνίες με τρίτες χώρες για την πολιτική συνεργασία αλλά και στο ζήτημα του ελευθέρου εμπορίου βλέπουμε, έχοντας ε, υπόψη την ε, υπογραφή της ΣΥΤΑ Νομίζω ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να ξεκινήσει, να αποτελέσει ένα έναυσμα για τις εμπορικές επαφές και σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες του ειρηνικού, όπως η Ιαπωνία και άλλες. Και νομίζω ότι θα αποστείλει μια ένα ισχυρό μήνυμα σε όλους εκείνους που αμφισβητούν και αμφιβάλλουν για τα ωφέλη της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς ε, θα ξεκινήσουν και οι διαπραγματεύσεις για το Brexit, υπάρχουν στη χώρα μου άνθρωποι που πιστεύουν ακόμη σε μια αγορά αυτοκρατορική και προ, υποστηρίζουν την, τις εμπορικές επαφές του Ηνωμένου Βεσσαλίου με χώρες της κοινοπολιτείας. Η αλήθεια όμως είναι ότι τώρα θα πρέπει να ε, επανεξεταστούν οι εμπορικές σχέσεις ε, υπό το φως της σύναψης ε, εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλες αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ πολύ και τώρα περνάμε στους Σκιώδης. Ξεκινούμε με, τον, με το ΕΛΚ, τον κύριο Ογκορίνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω και πάρα πολλά να προσθέσω μετά τις πολύ καλές παρατηρήσεις του κυρίου Τάνοκ. Να πω ότι είναι μια ξεκάθαρη έκθεση, δεν υπάρχουν επίμαχα θέματα. Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι η Νέα Ζηλανδία είναι ένας πολύ καλός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τις ίδιες αξίες, τα ίδια συμφέροντα, παρά την τεράστια γεωγραφική απόσταση που μας χωρίζει. Συμφωνία συνεργασίας για σχέσεις και συνεργασία με τη Νέα Ζηλανδία έρχεται ως επιβεβαίωση αυτών των εξαιρετικών σχέσεων, πολιτικών, οικονομικών σχέσεων στην έρευνα και την καινοτομία. Ο κύριος Τάνοκ, όπως αναμενόταν, έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ε, δεν βλέπω να υπάρχει καμία διαφωνία όσον αφορά την ε, τελική διατύπωση. Εμείς ε, προτιθέμεθα να καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες, αυτές όμως δεν θα αφορούν κάτι το συνταρακτικό και δεν θα διαταράξουν το πνεύμα που διαπνέει την έκθεση. Η Νέα Ζηλανδία ε, θα προχωρήσει σε μια συμφωνία ελεύθερων ανταλλαγών. Αυτό είναι και το επόμενο λογικό βήμα που θα ακολουθήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν βλέπω εκπρόσωπο των ε, σοσιαλιστών, ο κύριος Νικολάη. Ευχαριστώ εκ μέρους της Άλντε και εμείς ε, καλωσορίζουμε ε, κυρίως την προσέγγιση αυτού του ψηφίσματος που είναι ιδιαίτερα θετική. Έχουμε μια μακρά ιστορία που να αφορά στις ε, σχέσεις με τη Νέα Ζηλανδία και αναμφισβήτητα ε, συμμεριζόμεθα τις ε, ίδιες αξίες, δραστηριοποιούμεθα και οι δύο στα, στα, για τα ίδια θέματα και είναι γνωστό ότι η Νέα Ζηλανδία Ακόμα και είναι τόσο μακριά, η Νέα Ζηλανδία συμμετείχε σε διεθνείς σειράξεις όπως το Αφγανιστάν, Παραδείγματο χάρη. Τον Οκτώβρη είχαμε αυτή τη συμφωνία συνεργασίας, ε, μια πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό πολιτικό πλαίσιο για τις σχέσεις με τη Νέα Ζηλανδία. Η συμφωνία εξάλλου αφορά και θέματα αντιτρομοκρατίας, ε, τον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, κυρίως το κυβερνοέγκλημα στη Νέα ε, Ζηλανδία. Εκεί υπάρχει πάρα πολύ καλή εμπειρία. Περιμένουμε να υπάρξει μια νέα εμπορική συμφωνία γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εταίρος στην ανταλλαγή προϊόντων, άρα δηλαδή ήδη υπάρχουν πολύ καλές οικονομικές σχέσεις. Και κυρίως επιθυμούμε να καλωσορίσουμε την ε, τομεακή συνεργασία, τη γεωργία, την αλία, την ε, έρευνα, την τεχνολογία. Ε, θα καταθέσουμε κάποιες μικρές τροπολογίες, όχι δηλαδή κάτι που να απέχει κατά πολύ από την προσέγγιση του κυρίου Τάνοκ και ελπίζω ότι το ψήφισμα αυτό θα ολοκληρωθεί με πολιτική και νομική συμφωνία και θα αποτελεί μια πολύ καλή συνέχιση της συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νέα Ζηλανδία. Ευχαριστώ. Δεν έχω παρατηρήσει κάποιον άλλον να έχει ζητήσει το λόγο. Κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν είμαι σκιώδης και δεν θέλω να παρέμβω στη δουλειά των σκιωδών εισηγητών της ομάδας, αλλά θέλω να κάνω ε, τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, να ευχαριστώ τον εισηγητή για το ε, σχέδιο αυτής της έκθεσης να υπογραμμίσω κυρίως τα σημεία 3 και 4 όπου γίνεται λόγος για την Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορικών Ανταλλαγών για την εμπορική συνεργασία με τη Νέα Ισλανδία προφανώς αυτά έχουν σημασία στις διμερείς σχέσεις και πρέπει να παίξουν ρόλο και στις διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να δούμε ποιο νέο στοιχείο θα προκύψει, ποια θα είναι η διαφορά που θα προσθεθεί. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά το ποια θα είναι η μέσο μακροπρόθεσμη πρόπτικη και εμείς λοιπόν ενδέχεται να καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες και να δούμε λιγάκι την πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία με τη Νέα Ζηλανδία έτσι ώστε να εντοπίσουμε νέους τομείς ε, συνεργασίας ε, προς όφελος ε, της συνεργασίας, αμοιβαία συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισλανδία. Κύριε Τάνοκ, θέλετε και πάλι το λόγο. Να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε ότι χαιρετίζω τα σχόλια των συναδέλφων πολύ ευγενικά αυτά που είπαν κανένα πρόβλημα σε αυτή την έκθεση η σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισλανδία πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κλασικές, πολύ καλές σχέσεις με μια χώρα με την οποία έχουμε τις ίδιες αξίες κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα ε, και η προσέγγιση μας σε διεθνή θέματα ε, διεθνείς προκλήσεις όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη. Επίσης ε, και στην Ελληνικό, σε άλλες περιοχές. Παντού έχουμε τις απόψεις. Εγώ θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες, απλά και μόνο για την βελτίωση των σχέσεων και της φιλίας με αυτή τη χώρα που ναι με είναι πολύ μακριά, αλλά μας είναι πολύ οικία. Ε, πάρα πολλά πράγματα μαζί με μας. Αύριο είναι καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογίων και μετά θα τις εξετάσουμε στην συνάντηση των σκιωδών. The deadline is tomorrow at 11. Ευχαριστώ. Η προθεσμία υποβολή τροπολογιών αύριο 11 το πρωί. Και να πω ότι θα ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό στις 7 Σεπτεμβρίου. Επίσης, με ενημερώνει η Γραμματεία ότι το σημείο 7 θα αναβληθεί και θα συζητηθεί αύριο, καθώς ε, τα μέλη που συμμετείχαν στην αποστελή δεν κατάφεραν να είναι σήμερα εδώ, δεν θα καταφέρουν να είναι σήμερα εδώ στις 6. Οπότε με αυτά κηρύσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης. Συνεχίζουμε αύριο στις 9 το πρωί. Ευχαριστώ πολύ.